η γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, ειδικό έλεγχος Είναι εδώ η συγητής, ε, του δίνω λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στην έκθεση αυτή Μιλάμε για μια ανακοίνωση της Κομισιόν για την ε, γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα. Πρόκειται για τον, την οριοθέτηση αυτών των μειονεκτικών περιοχών. Πρέπει να βρούμε ένα νέο ορισμό. Αυτή τη στιγμή προσδιορίζονται με βάση κάποια εθνικά κριτήρια ποιες είναι αυτές οι μειονεκτικές περιοχές. Αυτά τα κριτήρια όμως είναι πολύ σημαντικά από κράτος σε κράτος. Δεν υπάρχει ομοιομορφία στα κριτήρια. Και το ελεκτικό συνέδριο έχει επικρίνει αυτή την ε, διασπορά. Τώρα η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της προτείνει ένα νέο τρόπο οριοθέτησης επί τη βάση οκτώ κριτηρίων. Αυτά τα κριτήρια θα μας οδηγήσουν σε μια όλος διόλου νέα χαρτογράφηση αυτών των περιοχών. Φυσικά δεν γνωρίζουμε από τώρα τις συνέπειες αυτών των κριτηρίων. Η Κομισιόν δεν έχει λάβει ακόμα τις προσωμιώσεις και δεν έχει ολοκληρωθεί ε, η διαδικασία. Τώρα, σε αυτή την έκθεση, εμείς τι προτείνουμε. Πιστεύουμε ότι ένας κοινό ορισμός είναι εκ των όνου κάνευ για να φτάσουμε σε μια ενιαία κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τη χρειαζόμαστε. Πιστεύουμε ότι οι αντισταθμίσεις και οι αποζημιώσεις που θα είναι η συνέπεια, η πιο σημαντική αυτής της νέας οριοθέτησης, Αυτές λοιπόν οι αντισταθμιστικές αποζημιώσεις είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, γεωργικής πολιτικής και θα μας επιτρέψει να προωθήσουμε τη γεωργία σε περιοχές που χωρίς αυτήν την αποζημίωση δεν θα υπήρχε δυνατότητα γεωργίας. Επίσης, ε, κάνουμε και μια αξιολόγηση των κριτηρίων. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτά τα κριτήρια θα λειτουργήσουν ή όχι, γιατί ακόμα που σας είπα δεν έχουμε τις προσωμιώσεις, δεν έχουμε όλα τα δεδομένα, αλλά Δεν νομίζουμε ότι αυτά τα κριτήρια επαρκούν. Θα πρέπει να δούμε επίσης αν τα κριτήρια που προτείνει η Κομισιόν θα παίξουν το ρόλο που θα ήθελε να παίξουν οι Κομισιόν. Αν θα τον παίξουν ατομικά ή αν θα πρέπει να συνδυάσουμε κάποια κριτήρια γιατί τα μειονεκτήματα συχνά οφείλονται σε περισσότερους από ένα παράγοντες. Μήπως θα πρέπει λοιπόν να συσσωρεύσουμε σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια κριτήρια. Επίσης, θα πρέπει να σκεφτούμε εάν θα πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή της επικουρικότητας. Χρειαζόμαστε νέα κριτήρια, χρειαζόμαστε ένα ευρύ πλαίσιο, όντω, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε και τη δυνατότητα στι χώρε και στι περιοχέ να κάνουν τι δικέ του μικροαλλαγέ και διορθώσει. Εν συνεχεία, η νέα αυτή χαρτογράφηση θα έχει την εξή συνέπεια ότι κάποιες χώρες δεν θα θεωρούνται πια ως μειονεκτικές περιοχές. Θα πρέπει για αυτές τις ε, περιπτώσεις, για αυτές τις χώρες και περιφέρειες να προβλέψουμε μια μεταβατική περίοδο. Επίσης, η ανακοίνωση της Κομισιόν πριν εφαρμοστεί θα πρέπει να τύχει κάποια επεξεργασία και θα πρέπει να ελέγξουμε πολύ συγκεκριμένα τις συνέπειες για τους γεωργούς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από το Κοινοβούλιο και κυρίως τους ε, υπεύθυνου και αυτούς που με βοήθησαν ε, για να συντάξω αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Είστε στο κατάλογό μου εξάλλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του έκθεση. Μιλάμε για τις μειονεκτικές περιφέρειες που είναι σημαντικό επιμέρους θέμα της ΚΑΠ αν θέλουμε να επιβιώσει η ΚΑΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει αυτές τις μειονεκτούσες περιοχές. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως τα κριτήρια είναι επαρκή και απολύτως κατάλληλα. Νομίζω ότι η Επιτροπή Γεωργίας θα πρέπει να αναδιατυπώσει αυτό το ζήτημα, διότι η Επιτροπή δεν μας έδωσε αποτελέσματα προσωμείωσης για τον ορισμό ενός φυσικού κριτηρίου. Γιατί αυτή η προσωμείωση δεν ήταν διαθέσιμη. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση προς την Κομισιόν. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει τόσο συχνά. Αν θέλουμε να αποτιμήσουμε τα πράγματα, θα πρέπει να έχουμε τα αποτελέσματα προσωμιώσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη από πλευράς Κομισιόν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να υπάρξει μια πρόταση κανονισμού και ελπίζω η Επιτροπή να λάβει υπόψη την έκθεση Dorfman και ελπίζω να μπορέσει να συνεχίσει τις εργασίες του επί του θέματος. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Äh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ σας ευχαριστώ για την ε, έκθεσή σας ε, κύριε Σιγητά. Λέτε ότι χρειάζονται ορισμένα επεξηγηματικά στοιχεία. Αυτό αληθεύει. Πιστεύω ότι το πλαίσιο το οποίο χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε αυτές τις ε, ε, περιφέρειες, τις περιοχές είναι πάρα πολύ ευρύ και χρειάζεται μια προσαρμογή. Υπάρχουν επίσης και τα κοινωνικά προβλήματα, δηλαδή ε, περιοχές που μειονεκτούν γιατί έχουν κοινωνικά προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα προβλήματα αυτά για την ύπαρξη την ίδια των περιοχών, την, ε, τις επιχειρήσεις τους. Χρειάζεται να καταρτιστεί λοιπόν ένας χάρτης με ειδικά κριτήρια για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των εκμεταλλεύσεων που έχουν ε, μία δυνατότητα επιβίωσης ή βιωσιμότητας. Υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες ε, στον γεωργικό τομέα, αλλά δεν θα πρέπει αυτά τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε να ε, ενισχύσουν αυτό το συνέστημα της αβεβαιότητας. Ευχαριστώ εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ. Βάσει της έκθεσης Dorfman, θα πρέπει το, ο προϋπολογισμός της ε, ΚΑΠ να καλύπτει τις ε, περιοχές που έχουν αυτά τα μειονεκτήματα. Αλλιώς θα υπάρξουν και κοινωνικά προβλήματα, αλλά και περιβαλλοντικά προβλήματα και καταστροφές. Καλωσορίζω λοιπόν την προσπάθεια της Κομισιόν που λέει ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ε, την ε, μήτρα των κριτηρίων. Σήμερα υπάρχουν διακρίσεις από κράτος μέλος σε κράτος μέλος ό,τι αφορά τις άμεσες πληρωμές, κάτι που είναι επιζήμιο κυρίως για τα νέα κράτη-μέλη, όπως τη Λετωνία, Φερρυπίν αλλά και άλλα νέα Στην Ουγγαρία το, η άρδευση ε, κάποιων αμοδών περιοχών είναι ιδιαίτερα προβληματική. Ε, υπάρχει μία απερίμωση αυτών των περιοχών. Θα πρέπει λοιπόν ε, το θέμα του νερού να το αντιμετωπίσουμε κατά προτεραιότητα. Ο monsieur le ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας κύριο Ντορφμάν και την εξαιρετική του εργασία σε αυτή την εισήγηση και νομίζω ότι ο τόνος της ερώτησής μου βασίζεται ε, στην έκθεση αυτή γιατί θέλω να απευθυνθώ στον ε, Επίτροπο, έχουμε αρχίσει αυτή την εργασία εδώ και πολλούς μήνες, δημιουργούνται αντιδράσεις έντονες σε διάφορες χώρες οι οποίες θα χάσουν το καθεστώς που έχουν αυτή τη στιγμή ε, των, της, ε, των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα και αυτό παρεμβαίνει σε μια χρονική στιγμή όπου υπάρχουν δυσκολίες για ορισμένες παραγωγές και για ορισμένες περιοχές. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε γρήγορα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τρία ολόκληρα ολόκληρα χρόνια πριν να έρθει μια σαφής απάντηση που να, για αυτούς τους γεωργούς που έχουν το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Εσαϊά. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με το γεγονός ότι οι περιοχές που μειονεκτούν αποτελούν το επίκεντρο αυτής της έκθεσης. Βεβαίως ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε μια βιώσιμη γεωργία και για το μέλλον της Ευρώπης. Θα πρέπει να ορίσουμε επαρκή ε, κριτήρια, ε, γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Ιδιαίτερα ως προς τη γεωργία στις μειονεκτούσες περιοχές. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι προγενέστερες μεταρρυθμίσεις ε, δεν κάλυψαν τις ανάγκες αυτών των περιοχών και θα πρέπει να μπορέσουν αυτές οι περιοχές να, να μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγή τους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε επαρκή κριτήρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα κατάφερε πολύ καλά με τις ε, γαλακτοκομικές ποσοστώσεις, ιδιαίτερα όταν δεν τις έλαβε υπόψη. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις διαφορετικές γεωργικές ε, συνθήκες, τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, εδαφικές συνθήκες, καθώς και ιστορικές ε, και κοινωνικές ε, παραμέτρους. Όλες αυτές οι προαναφερθήσεις περιπτώσεις επηρεάζουν την παραγωγή και τις οικονομικές επιδόσεις. Σημερίζομαι την ανησυχία του εισηγητή για την καταλληλότητα των κριτηρίων. Χρειαζόμαστε μια πιο ενδελεχή ανάλυση. Πρέπει να κάνουμε επίσης και μια μελέτη αντικτύπου. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτές τις περιοχές υπό την κοινή αγροτική πολιτική. Και πρέπει να τις υποστηρίζουμε στο σωστό επίπεδο. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, ευχαριστώ τον κύριο Ντόρφμαν για τη θαυμάσια έκθεση για την ανακοίνωση της Κομισιόν για μια καλύτερη στοχοθέτηση της ε, βοήθειας προς τους ε, αγρότες ε, σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα. Ο συνολικός στόχος των πληρωμών αυτών σε τέτοιες περιοχές είναι να εξασφαλίσουμε τη χρήση της γεωργικής γης και να διατηρήσουμε την ύπεθρο ως έχει καθώς και τα βιώσιμα γεωργικά συστήματα. Ε, τα, οι πληρωμές αυτές ε, αντισταθμίζουν το επιπλέον κόστος για τους γεωργούς και την απώλεια εισοδήματος ε, λόγω των φυσικών μειονεκτημάτων των περιοχών τους. Το Συμφούλιο αποφάσισε να διαγράψει από τους στόχους τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Η διαγραφή των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων θα πρέπει να θεωρηθεί μέσα στο πλαίσιο του συνόλου των μέτρων που είναι στη διάθεση των κρατών μελών στα πλαίσια του κανονισμού ε, για την Ήπεθρο, ε, για την ανάπτυξη των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των τουριστικών δραστηριοτήτων και την παροχή βασικών υπηρεσιών κτλ. Επομένως, οι πληρωμές για τα φυσικά μειονεκτήματα δεν γίνονται για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της μείωσης του πληθυσμού. Το να πληρώνουμε τους γεωργούς σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για την παραγωγή τους θα στρεβλώσει τον ανταγωνισμό με γεωργούς σε άλλες περιοχές. Επίσης, η κοινωνική και οι οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτε αλλάζουν συν χρόνο. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται μια παρακολούθηση και μια αναθεώρηση τη κάθε περιοχή. Η πρόταση για να λάβουμε υπόψη την, το απόμακρο των περιοχών αυτών δεν είναι κατάλληλη. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακότητα, υπάρχουν και άλλοι τρόποι προσδιορισμού. Παραδείγματο χάρη το άρθρο για το ειδικό, τα ειδικά μειονεκτήματα του, που αναφέρει ο κανονισμός. Η Κομισιόν έχει καλέσει τα κράτη-μέλη ούτως ή να υποβάλουν εναλλακτικέ προτάσεις για τα φυσικά κριτήρια και τα κατόφλια τους. Αυτές οι προτάσεις θα αναλυθούν από τους επιστήμονες, ε, θα δούμε κατά πόσον ισχύουν και θα δούμε αν είναι διαφανή αυτά τα κριτήρια και αν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε σωστά. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Θα πρέπει να τεστάρουμε το, την οριοθέτηση. Και η Κομισιόν μετά το 2013 ε, θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα. Εκείνες οι περιοχές που μπορεί να χάσουν το καθεστώς τους, θα, για αυτές τις περιοχές θα προβλεφθεί ε, μία ειδική περίοδος μετάβασης. Ευχαριστώ, Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος. Τελειώνει η συζήτηση. Θα ψηφίσουμε για το σημείο αυτό σε δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες, στην ε, Μίνιο Ολομέλεια.